ενημερωτικό υλικό στους ασθενείς. Είναι πάντοτε ευθύνη των γιατρών και εδώ εμείς δεν πρέπει να παρέμβουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώθηκε εκείνη η συζήτηση. Η πληροφορία θα γίνει την Τετάρτη στις 12. L'ordine την, ε, με βάση τη σημερινή διάταξη προχωρούμε στην έκθεση Evans, περιορισμό τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ξεκινούμε τη συζήτηση. Δίνοντα το λόγο στον εισηγητή για τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ κύριε εισηγητά. Thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου που κατέστησαν δυνατή αυτή τη συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όλου του σκιώδει εισηγητέ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ισπανική και τη Βελγική Προεδρία, καθώ και την Επιτροπή Περιβάλλοντο ε, και το προσωπικό και του βοηθού στην ομάδα. Κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία μετά από σκληρή και επικοδομητική δουλειά η οποία περιλάμβανε και δύσκολες συμβιβαστικές λύσεις. Πάνω από 9 εκατομμύρια τόνοι ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πολλούνται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μεγάλο μέρος αυτών είναι οικιακός εξοπλισμός ε, και εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ε, και ε, οικιακών συσκευών. Όσο αυξάνεται η αγορά, σιγά σιγά θα γίνει μια πηγή αποβλήτων που θα φτάσει στα 12,3 τόνους το 2020 είναι πολύπλοκα υλικά και περιλαμβάνουν πολλές επικίνδυνες ουσίες. Είναι λοιπόν σημαντική προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στις επικίνδυνες ουσίες, ε, ιδίως σε ουσίες που εμποδίζουν την ανακύκλωση ή δημιουργούν κινδύνους για το περιβάλλον κατά την ε, μεταποίησή τους. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η τρέχουσα οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ροζ δηλαδή, έχει εμποδίσει διάφορες κατηγορίες υλικών όπως τα επιβραδυτικά φλόγας να φτάνουν στην ανακύκλωση. Η οδηγία ΡΟΣ έχει θέσει λοιπόν υψηλά πρότυπα, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια και με την αναδιατύπωση χρειάζεται ιδιαίτερη ανάληψη ευθύνη, ούτω ώστε να είναι πιο φιλόδοξη η νομοθεσία που θα υιοθετήσουμε. Νομίζω ότι έχουμε βελτιώσει την τρέχουσα οδηγία ποικιλό τρόπο. Τώρα Υπάρχει σαφής μεθοδολογία με κριτήρια ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις για νέους περιορισμούς ανεξάρτητα από τη ΡΙΤΣ και συμπληρωματικά προς τη ΡΙΤΣ. Έχει επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή για να συμπεριλαμβάνονται όλα, όλοι οι ηλεκτρικοί και ηλεκτρονικοί εξοπλισμοί μέσα στα επόμενα χρόνια, εκτό αν ε, δίδεται ρητή εξαίρεση. Θα υπάρχουν ε, ε, σαφεί εξαιρεσει για τρία χρόνια και καθώ και εξέταση φθαλικών προϊόντων και προϊόντων επιβραδυτικών φλόγας, τα οποία έχουν οριστεί ως προτεραιότητα. Με βάση σαφή κριτήρια και σαφείς χρονικές προθεσμίες θα δοθούν οι εξαιρέσεις, θα εξεταστούν και τα νανοηλικά πολύ συγκεκριμένα ε, σε μελλοντική αξιολόγηση. Είναι πολύ φιλόδοξη αυτή η έκθεση και δεν θα ε, σας εκπλήξω αγαπητοί συνάδελφοι να σας πω ότι δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένη με το τελικό αποτέλεσμα. Η οδηγία ΡΟΣ ήθελε να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα συγκεκριμένων αποβλήτων και νομίζω ότι χάσαμε μία ευκαιρία να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προσθέτοντας επιπλέον περιορισμούς. Όμω έχουμε κρατήσει τη βασική ταυτότητα τη οδηγία και έχουμε ενδυναμώσει την πρόταση τη επιτροπή ε, σε πολλού τομεί. Για τους πίνακε συσχέτιση, Εμεί πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί για τα κράτη-μέλη, αλλά αυτό είναι ένα οριζόντιο θέμα το οποίο έχει επίπτωση στο σύνολο τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και δεν μπορεί να επιληθεί σε αυτό το φάκελο, σε αυτό το θέμα και μόνο. Για να μπορέσουμε να βρούμε μία λύση, στην Ατροπολογία 105 πρότεινα να έχουμε μία δήλωση που θα ζητάει από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για την πρακτική των κρατών μελών όσον αφορά τους πίνακες συσχετισμού και, αυτό, ε, και το κατά πόσο αυτό επηρεάζει τη δουλειά της Επιτροπής. Αυτό θα μας δίνει μια σαφέστερη εικόνα για τη μελλοντική συζήτηση. Πιστεύω ότι μία όριστη και μη φιλόδοξη πρόταση καταφέραμε με τις τροπολογίες μας να την κάνουμε φιλόδοξη πρόταση που θα βοηθήσει το περιβάλλον και τώρα και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Δαμανάκη έχει το λόγο ξενόματος επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο υπεύθυνο επίτροπο, κύριο Ποτότσικ είναι εδώ μαζί μου, αλλά δυστυχώ θα σιωπά, διότι έχει ένα πρόβλημα στο λαιμό του. Δουλεύει επιμακρών για το θέμα αυτό και θα λειτουργήσω ως φωνή του. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι και κυρίε βουλευτέ. Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση για την αδιατύπωση τη οδηγία για του περιορισμού επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Πρέπει να πω ότι δεν θα είχαμε πετύχει, δεν είχαμε φτάσει στο σημείο αυτό αν δεν υπήρχε η σκληρή δουλειά του Κοινοβουλίου στο πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή την εισηγήτρια κυρία Evans και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας ε, Τροφίμων για την εξαιρετική δουλειά που διεξήχθη για το θέμα αυτό. Από την είδηση της, το, κείμενο, το νομοθετικό κείμενο ήταν επιτυχές. Ε, απέφυγε ε, χιλιάδες τόνους κακών ουσιών από διάθεση και ε, να, την απελεπιθανή απελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Έφερε σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό ηλεκτρονικών προϊόντων ε, στην Ένωση αλλά και παγκόσμια. Άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η μεγάλη εμπορική εταιρεία της Ένωσης, ακολούθησαν τα παραδείγματα της Ένωσης, προωθώντας παρόμοια νομοθεσία χρησιμοποιούμε τεράστιους όγκους ηλεκτρονικών προϊόντων και που αυξάνονται και περιλαμβάνουν πολλέ πολλές επικίνδυνες ουσίες. Ένας κομπιούτερ περιλαμβάνει πάνω από 60 πρώτες ύλε. Κατά μέσο όρο, κάθε πολίτης της Ένωσης παράγει 25 κιλά ηλεκτρονικών αποβλήτων το χρόνο. Ο νόμο, η νομοθεσία αυτή θα εξασφαλίσει ότι τα ηλεκτρονικά προϊόντα δεν θα έχουν πλέον πολλέ επικίνδυνε ουσίε και θα διευκολύνει την ανακύκλωση των ε, προϊόντων αυτών. Άρα συμβάλλει και στην ε, μετατροπή της Ένωσης σε πιο αποτελεσματική, αποτελεσματικό χώρο στη διαχείριση των πόρων. Ωστόσο, ο κλάδος και τα κράτη-μέλη αναφέρθηκαν στον κίνδυνο ανεπαρκούς ή μη ε, ενδεδειγμένης εφαρμογής οδηγίες. Το status quo, ωστόσο, είναι ανεπαρκέ όχι μόνο σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντο αλλά και τη δημιουργία ε, ισότιμης αντιμετώπιση στο εσωτερικό τη Ένωση. Γι' αυτό είναι σημαντικό η νομοθεσία αυτή να διευκρινιστεί και να απλουστευτεί. Το βασικό στοιχείο για την Επιτροπή είναι να, να εξασφαλιστεί η προσέγγιση με το REACH προ όφελο τα, τα πραγματικά περιβαλλοντικά ωφέλη υλοποιούνται μόνο όταν εφαρμόζονται σωστά οι νόμοι σε εθνικό επίπεδο. Ελπίζω ότι η εισαγωγή των κοινών ορισμών και των εργαλείων αξιολόγηση στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, για την πρόθεση στην αγορά των, εμπόδι, προϊόντων θα βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση. Επιπλέον, η περιβαλλοντική στόχοι της οδηγίας βελτιώνονται μέσω της επέκτασης της κάλυψης προϊόντων Πρώτον, στι δύο νέε κατηγορίε, ιατρικά εργαλεία και εργαλεία παρακολούθηση και ελέγχου και σε 8 χρόνια των ε, διπλών ηλεκτρονικών προϊόντων. Η, η περαιτέρω επέκταση του πεδίου εφαρμογή τη νομοθεσία αυτή θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο τα οικονομικά κέρδη, αλλά οι οικονομικοί φορεί θα πρέπει προφανώ να έχουν επαρκή χρόνο για να προσαρμοστούν και οι αλλαγέ να γίνονται πάντα με βάση στέρη ενημέρωση. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή θα προχωρήσει σε αναθεώρηση του πεδίου εφαρμογή σε σχέση με την υφιστάμενη νομοθεσία, που δεν έχει αποκτήσει ακόμα αξιολόγηση αντικτύπου. Θέλουμε να διευκρινίσουμε λοιπόν το θέμα με δύο δηλώσει. Πρώτον, για το πεδίο εφαρμογή. Η Επιτροπή ερμηνεύει το κείμενο ότι βάσει του άρθρου 2α, 2.1α διορθώνει μιλήτρια, Κατά τη διάρκεια τη μεταβατική περίοδου μέχρι τα 8 έτη, τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να επιτρέψουν στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα που ήταν εκτός του πεδίου εφαρμογή τη Οδηγία 95 του 2002, αλλά που θα υπαχθούν στη νέα οδηγία, να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά του. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση, βάσει του άρθρου 19, α, η Επιτροπή προτίθεται να αναλάβει το αργότερο τρία έτη μετά τη θέση ισχύ της ε, παρούσης οδηγίας αξιολόγηση αντικτύπου με έμφαση στις αλλαγές στο πεδίο εφαρμογή. Η αναθεώρηση αυτή μπορεί να οδηγήσει στην υποβολή από πλευρά Επιτροπή νέα νομοθετική προτάσεω βάσει του δικαιώματο νομοθετική πρωτοβουλία που διαθέτει βάση των συνθήκων. Επίση, θέλουμε να, να προβούμε στην ακόλουθη δήλωση για τα νέα υλικά. Ξέρουμε ότι οι εργασίε προ τον κοινό ορισμό των, ε, του υλικού αυτού συνεχίζεται στην Επιτροπή. Θέλουμε να προδιοθετήσουμε μια σύσταση για αυτόν τον κοινό ορισμό για, κάθε, ε, για όλο τον κλάδο, τον νομοθετικό κλάδο στο εγγύ μέλλον. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πρόταση ΡΟΣ καλύπτει διάφορες πηγές και νανοπηγές των ουσιών των ενώσεων αυτών που απαγορεύονται και που θα υπαρχθούν σε, με, σε κατά προτεραιότητα αναθεώρηση. Τέλος, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για την έλλειψη υποστήριξης στη διάταξη που υπήρχε στην πρώτη της Επιτροπής και που καθιστούσε την θέσπιση πινάκων στις υποχρεωτικών. Δεχόμαστε την ε, υποκατάσταση της διάταξη από μια αιτιολογική σκέψη που θα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν την πρακτική αυτή για να διευκολυνθεί μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Δηλώνουμε ωστόσο ότι τούτο δεν πρέπει να θεωρηθεί ως προηγούμενο. Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε οριζόντια λύση με, το, με τα συνομοθετικά όργανα σε αυτό το ζήτημα. Η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί το πακέτο συμβιβασμού για να επιτευχθεί συμφωνία στην οδηγία σε πρώτη ανάγνωση θα ζητούσαμε και από το Κοινοβούλιο να θετήσει την ίδια θέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξεκινούμε τις συζητήσεις με τους αγωγητές από τις πολιτικές ομάδες. Ξεκινούμε με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο κύριος Σόνικ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Evans, γιατί είναι πολύ καλή η δουλειά που έκανε στον τομέα αυτό. Χωρί την δική της δέσμευση δεν θα καταλήγαμε σε συμβιβαστικές λύσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων στην πρώτη ανάγνωση. Η οδηγία ΡΟΣ μιλά για το περιβάλλον, μιλά για την ανάπτυξη και προσπαθήσαμε να μειώσουμε τα απόβλητα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ε, εξοπλισμών. Κατά την αναδιατύπωση της οδηγίας, ε, προτεραιότητά μας ήταν η θέσπιση πιο υψηλών προτύπων. Η νέα οδηγία θα οδηγήσει όλους τους κατασκευαστές ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο να προσαρμοστούν με τα νέα πρότυπα και προδιαγραφές και είναι κάτι το οποίο θα δώσει σωστές κατευθύνσεις και στους κατασκευαστές. Είναι πολύ καλές οι συμβαστικές λύσεις στις οποίες έχουμε καταλήξει. Η νέα οδηγία, η νέα οδηγία ΡΟΣ δίνει επαρκή χρόνο προσαρμογής στους κατασκευαστές. Η προτινόμενη μεθοδολογία βασίζεται στη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε με την REACH και θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Λέινεν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω ότι θα ξαναβρει γρήγορα την φωνή του Επίτροπο, γιατί χρειαζόμαστε τη φωνή του στη διάσκεψη για το κλίμα στην Κανκούν. Και μετά την αναθεώρηση τη Αλία, μου κάνει εντύπωση που η κυρία Δαμανάκη έμεινε και για την, έμεινε και για την αναδιατύπωση τη οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού. Ευχαριστούμε πολύ που μα κάνετε τη τιμή. Είναι κρίμα που λείπει το παράρτημα 3. Κρατάμε όμως τις ε, ουσίες αυτές ε, κατά και κατά την αναθεώρηση μετά από τρία χρόνια θα γίνει η αξιολόγηση επιπτώσεων ε, και θα εξετάσουμε αν ουσία τι προβλήματα υπάρχουν. Υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις και θα πρέπει να εξετάσουμε ε, τι κενά υπάρχουν, τι ελλείψεις υπάρχουν που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα για την ανθρώπινη υγεία. Όπως ε, με ε, το κάδμιο που περνάει στο περιβάλλον μέσω των ηλιακών συσσωρευτών. Ε, ελπίζουμε ότι ε, η σημαντική αυτή πρόοδος θα συνοδευτεί από περαιτέρω πρόοδο τρία χρόνια αργότερα κατά την ε, επανεξέταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και του σκιώδη συζητητές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κράμερ, εκ μέρου της ομάδα Άλντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, με την οδηγία αυτή ε, εκπλήσωμε διότι καταλήξαμε σε τόσο γρήγορη συμβαστική λύση. Είναι μια συμβαστική λύση την οποία θεωρούμε εφικτή. Είναι δύσκολος ο δρόμος που ακολούθησε αυτό το νομοθετικό κείμενο στο Κοινοβούλιο. Ε, προσπαθήσαμε κάποιες ουσίες ε, να τις ορίσουμε ως ιδιαίτερα επικίνδυνες, το PVC, τα νανοηλικά, ουσίες τις οποίες αποκαλέσαμε ε, επικίνδυνες που δεν θεωρήσαμε τελικά σκόπιμο να κρατήσουμε αυτόν τον ορισμό. Είναι πολλοί οι συμβασμοί λοιπόν τις οποίες, ε, τους οποίους κάναμε. Και προσπαθήσαμε ε, να ακολουθήσουμε ιδιαίτερα ορθολογική κατεύθυνση στις συζητήσεις μας. δεν μπορούμε εξαφνικά ε, να περάσουμε στην πλήρη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, ιδιαίτερα με, για τον τομέα της ενέργειας. Ελπίζουμε ότι στα απόβλητα των ηλεκτρονικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών δεν θα συμβούν τα ίδια τα οποία συνέβησαν στον τομέα της ενέργειας, γιατί θα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ευχαριστώ πολύ. Για την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, η κυρία Γκέρλινγκ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή και του συνεργάτε του. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις ε, πέσαμε σε μια συμφωνία που μπορούμε να την προσυπογράψουμε. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ με την ευκαιρία αυτή σε κάποιους τομείς. Αυτή η αναδιατύπωση σκοπό είχε να βελτιώσει εξορισμού την κατάσταση. Έτσι κάνουν οι αναδιατυπώσεις σκοπό είχε να, εξα... απλουστεύσει τις απαιτήσει ε, από τους κατασκευαστές. Θεωρώ ότι κάνουμε ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω σε πολλούς τομείς. Είναι ευπρόσεκτο το παράρτημα 3 που είναι μαύρος κατάλογος για πολλές ουσίες, αλλά δυστυχώς λυπάμαι τη διαθεσιμότητα των κριτηρίων, ως κριτήριο μάλλον. Επίσης, δημιουργήθηκε για την ύπαρξη νομικής ασφάλειας θέλω να αφαιρθώ στο σημείο εφαρμογής. Εγώ από την αρχή υποστήριζα ότι θα υπάρξει περαιτέρω έλλειψη νομικής ε, ε, ε, ασφάλειας λόγω της, των αιτήσεων για πολλές εξαιρέσεις. Τώρα, οι έλεγχοι που υπάρχουν στον κανονισμό θα δημιουργήσουν κάποια προβλήματα και είναι πρόσδεκτη η αφοσίωση και η δέσμευση της Κομισιόν να τα μελετήσει εκ των υστέρων, αλλά ίσως θα ήταν καλύτερα να τα είχε κάνει από πριν. Διερωτώ με πώς αυτή η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή έχει ε, προωθήσει και την ε, σαφήνεια αλλά και την νομική ασφάλεια. Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω το κίνδυνο υπερβολικών κανονισμών Υπάρχει και η οδηγία για τις χημικές ουσίες, για τις επικίνδυνες ουσίες, υπάρχουν οι κανονισμοί REACH και η εφαρμογή τους εξελίσσεται και όπως ακούσα από την Κομισιόν ικανοποιητικά. Κάποια στιγμή πρέπει να αφήσουμε το REACH να μας καθοδηγήσει όπως ακριβώς πρόκειται να γίνει. Θέλω όλα αυτά να τα λάβει υπόψη της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ομάδα GUE. Το λόγο έχει η κυρία Βίλς για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια διότι έκανε εξαιρετική δουλειά και παρότι υπήρχε μεγάλη αντίδραση από το Συμβούλιο και από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου καταλήξαμε σε αυτό το πολύ θετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτή η πρόοδο ε, ε, πραγματικά ε, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο. Αυτό που είναι αρνητικό είναι ότι ο κατάλογο των απαγορευμένων μέχρι τώρα ουσιών, που ήταν έξι μέχρι τώρα, έχει επεκταθεί με θελικές και άλλες ουσίες. Από αυτές τις ουσίες τίθενται σημαντική κίνδυνη και δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ήδη από τη θέση εφαρμογή το 2011 ένας κατασκευαστής θέτει σε εμπορία κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς υπολογιστέ ε, χωρίς ε, τα, τις ε, επιβλαβείς αυτές ουσίες και χωρίς να αυξάνεται το κόστος παραγωγής. Νομίζω ότι εγκαταλείψαμε μια ευκαιρία να κάνουμε την βιομηχανία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών λίγο πιο φιλική προς το περιβάλλον θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τις εταιρείες ε, για να κάνουν τις σημαντικές προόδους που είναι απαραίτητες. Κάθε χρόνο ε, εκατομμύρια τόνων αποβλήτων επιβαρύνουν το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι προς εις βάρος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. για την ομάδα EFD, ο κύριος Ρώση για ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι, εμείς εκφραστήκαμε κατά της πρώτας οδηγίας, πολύ έντονα και στην Επιτροπή, διότι ο, η συγγήτρια έκανε τεράστιες τροπολογίες, τροποποίησης των προτάσεων της Κομισιόν, άλλαξε το πεδίο εφαρμογή και είπε ότι πρέπει να καταργηθούν άλλες 33 ουσίες στο παράρτημα 3, μεταξύ των οποίων και οι επιβραδυντές φλόγας, PVC και πολλές άλλες. Και επίσης μείωσε τις ε, περιόδους χάριτος και τις εξαιρέσεις και έβαλε αυστηρότερους κανόνες στα νανοηλικά αυτά τα οποία δεν στηρίζονται από επιστημονικά στοιχεία και αν εγκριθούν από την Ολομέλεια θα επηρεάσουν σημαντικά τις επιχειρήσεις και τις ε, θέσεις εργασίες. Ευτυχώς χάρη στον τριμερή διάλογο και χάρη στους ε, σκιώδεις εισηγητές καταλήξαμε σε, κάποια, ε, σε κάποιο συμβιβασμό και την ανάγκη αναθεώρησε τρία χρόνια. Ένα άλλο επικίνδυνο σημείο ήταν τα ανανοηλικά. Το κείμενο τροποποιήθηκε από τροπολογίες και στον τριμερή διάλογο καταλήξαμε σε ένα ε, πού μπορούμε να στηρίξουμε. Άλλοι ομιλητές ε, τώρα, η κυρία Βάσκερ. Κυρία Βάσκη, έπρεπε λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η οδηγία ΡΟΣ είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Υπάρχουν ε, πολλά τα οποία δημιουργούν διαφορές και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα ε, για το καλό αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε μετά τις τριμερείς συζητήσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριμένα σημεία. Καταρχήν, το πεδίο εφαρμογή, Για ποιο εξοπλισμό θα πρέπει να ισχύσει αυτή η οδηγία. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αρχικά το πεδίο εφαρμογή αφορούσε οικιακό εξοπλισμό, λευκές συσκευέ οικιακή χρήση. Υπάρχουν πολλά προϊόντα και λόγω της χρήσης νέων τεχνολογιών. Ο στόχος της οδηγίας ήταν διαφορετικά, διαφορετικός αρχικά. Θα έπρεπε να είναι πολύ υψηλότερα τα πρότυπα προστασίας για τον οικιακό εξοπλισμό από ότι για το τεχνολογικό εξοπλισμό που εγκαθίσταται από ειδικό προσωπικό και στη συνέχεια ανακυκλώνεται κλπ. δεν ήμουν υπέρ της αλλαγής στο πεδίο εφαρμογή, αλλά είδα ότι η πλειοψηφία ήθελε αυτή την ε, κατεύθυνση. Δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικό μειονέκτημα και γι' αυτό καταλήξαμε σε αυτή την πρόταση και για το παράρτημα 3. Άλλε 23 ουσίε θεωρήσαμε σκόπιμο να θεωρηθούν ουσίε προτεραιότητα ούτως ώστε να καταλήξουμε τελικά ε, σε ε, απαγόρευση. Χαίρομαι για το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε μετά από τις συζητήσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Βαν Μπρέμπτ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας την κυρία Εύεν στην συγκήτρια. Έδειξε πραγματικά εξαιρετικά αποφασιστικό χαρακτήρα ε, στην επίτευξη του αποτελέσματος αυτού που μπορούμε να υποστηρίξουμε διότι συνιστά πραγματική βελτίωση. Περιέχει πολλά καινούργια θετικά στοιχεία Μερικά από τα οποία σχετίζονται με την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή. Καλύτερα θα ήταν να έχει γίνει νωρίτερα αυτό, αλλά καλή αργά παρά Υπάρχει μια οδηγία που είναι ανεξάρτητη από το REACH, ακόμα και τώρα, παρότι υπάρχουν οι πίνακες αντιστοιχίες. Πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό πως πετύχαμε μια καλή συμφωνία στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αναθεωρήσουμε τις συνέπειες των χημικών ε, ουσιών στο μέλλον. Υπάρχουν άλλα προϊόντα, τα HCBBD, αν τα προφέρω σωστά, που είναι οι επιβραδυντές καύσεως ε, που αποτελούν προτεραιότητα. Επίσης πρέπει να ληφθούν ε, μέτρα για τα προϊόντα. Θέλουμε να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, μια και θα κάνει δήλωση η Επιτροπή, θεωρώ κάτι, ότι είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν και άλλες ε, πτυχές ε, που δεν μας ικανοποιούν βέβαια. Σαν πολιτική ομάδα θα θέλαμε να υπάρχουν και κάποιες άλλες έξω χημικέ ουσίες, να υπάρχει ταχύτητα για να θεωρήσει ε, μικρότερος αριθμός εξαιρέσεων. Μια τελευταία παρατήρηση, χρειάζεται να επανέλθω στο θέμα των ε, ηλιακών πάνελ. Οι σοσιαλιστές ήταν η μόνη ομάδα που μέχρι την τελευταία στιγμή ε, είχαν αμφισβητήσει την το να εξαιρεθούν τα πάνελ από την οδηγία. Κάτι που θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο για τα επόμενα δέκα χρόνια το κάνδμιο που μετά το 2003 απογοητεύτηκε θα παραμείνει σε κυκλοφορία. Αυτό είναι κρίμα. Κρίμα για έναν κλάδο που θα έπρεπε να, να παίζει ε, ηγετικό ρόλο και να είναι παράδειγμα. Ωστόσο η ομάδα μου θα υποστηρίξει με ικανοποίηση τη συμβαστική λύση ε, και Ελπίζω να μην έχουν λάθος ενημέρωση η ομάδα EFD γιατί δεν τους είδε στον τριμερή διάλογο. Ο κύριος Νέλχαρτ για ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, με την αναδιατύπωση της οδηγίας θέλουμε να συνεισφέρουμε στην προστασία του καταναλωτού και τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει γιατί θέσαμε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, ένα πλαίσιο που είναι καλό και για τους καταναλωτές και για το περιβάλλον, αλλά θα δίνει και ασφάλεια στις επιχειρήσεις για επενδύσεις ε, και για καινοτομία. Αυτό και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να επεκταθούν στον τομέα της έρευνας. Και αυτό ε, είναι για μας καθησυχαστικό και είναι κάτι το οποίο μας οδήγησε στην ε, συμφωνία μας τελικά ώστε να έχουμε ε, μια κοινή θέση. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια ακούσαμε ότι πολλοί συνάδελφοι είπαν ότι ε, ε, λυπούνται γιατί τα ηλιακά πάνελ δεν ε, συμπεριλαμβάνονται. Μιλάμε για το κάδμιο. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και υπάρχει μια μεγάλη διαφορά γιατί δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα μαζί και να πούμε ότι οτιδήποτε ε, είναι επιζήμιο θα το απαγορεύσουμε. Θα μπορούσαμε να απαγορεύσουμε και το θιάφι σε άλλες ε, ε, χρήσεις. Αλλά τώρα έπρεπε να περιοριστούμε στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Και όσον αφορά το PVC, οι εταιρείες οι οποίες παράγουν το PVC πρέπει να προσαρμόζουν τη τεχνολογία τους στις νέες απαιτήσει. Εγώ είμαι ικανοποιημένος με αυτά τα οποία έχουμε τώρα ενώπιόν μα. Πιστεύω ότι με αυτό μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε πολλά και για τους καταναλωτές και για το περιβάλλον και για την καινοτομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τεταρέλα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια διαπιστώσαμε μεγάλε προσπάθειε των κοινοτικών οργάνων με στόχο να καταστήσουν την παρασκευή χρήση και διάθεση των ηλεκτρονικών προϊόντων με μεγαλύτερο σεβασμό προ το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η οδηγία Ρότχα είναι ένα, μια ψηφίδα στην πολιτική αυτή. Η συμφώνηση με την οδηγία αποτελεί ωστόσο μια τεράστια πρόκληση για τι επιχειρήσει, αλλά και ευκαιρία ταυτόχρονα διότι η ικανότητα να παράσχουν προϊόντα που ρηπαίνουν λιγότερο γίνεται ε, ένα βασικό στοιχείο διαφοροποίησης των επιχειρήσεών μας που είναι πολύ σημαντικό και τέτοιο που να αποκτά ένα πραγματικά χαρακτήρα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Δεν πρέπει οι επιχειρήσεις να βλέπουν ε, τις διατάξεις οδηγίες υποχρεωτικά ή ε, κάτι το υποχρεωτικό και προβληματικό, αλλά μια ευκαιρία προώθηση των προϊόντων τους. Ε, κάποιες ωστόσο εξαιρέσεις ε, είναι αναγκαίες, που οφείλονται και στην υφιστάμενη κρίση ή γιατί θα εξεταστούν από μεταγενέστερη οδηγία. Τα νάνο προϊόντα, το ζήτημα ασφάλειας, οι πάγιες εγκαταστάσεις, τα, τα μηχανήματα μετακίνησης, οι ιατρικά εργαλεία, τα φωτοβολταϊκά πάνελ και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για έρευνα και ανάπτυξη. Με την ίδια ευκαιρία θέλω να ευχηθώ να υπάρχει μια μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ της παρούσης οδηγίας και του κανονισμού REACH, αποφεύγοντας οποιαδήποτε περίπτωση σύγχυσης ή επικάλυψης, διότι και οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις χρειάζονται σαφείς κανόνες. Ευχαριστώ. Το λόγο έχουν τώρα οι αγωγητές ε, μέσω της διαδικασίας Catch the Eye. Ξεκινούμε από τον κύριο ER. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να υποστηρίζουμε την οδηγία αυτή Πιστεύουμε ότι η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στις απαιτήσει που υπήρχαν. Παραμένουν βέβαια κάποια μικρά θέματα τα οποία θα έπρεπε να συζητηθούν περαιτέρω. Σε όλα όσα κάνουμε θα πρέπει να έχουμε κατά νου τη διεθνή διάσταση δεν είναι επαρκές ε, το να παραμένουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, καθαροί από τέτοιες ουσίες αλλά να επιτρέπουμε εισαγωγές τέτοιων ουσιών στα προϊόντα μας. Χρειαζόμαστε σαφείς διατάξεις ε, και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και τις τα γραφειοκρατικά προβλήματα. Και τρίτον, θα πρέπει η διαδικασία αυτή να είναι δυναμική και όχι στατική και γι' αυτό χρειαζόμαστε τακτικά επανεξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, είναι ένα μικρό βήμα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η τροποποίηση που έχουμε ενώπιόν μας συμπεριλαμβάνονται όλε οι ουσίε μαζί και οι εξαιρεσει τι οποίε έχουμε συμπεριλάβει και νομίζω ότι δίνουν μια σαφή κατεύθυνση στον κλάδο. Αυτό που είναι σημαντικό για την οδηγία είναι η ενημέρωση των καταναλωτών. Είναι πολύ σημαντικό για την οδηγία αυτή για τα απόβλητα ηλεκτρονικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού να γνωρίζουν οι καταναλωτές ε, ποια είναι, ε, τα, ε, ποιοι είναι οι ρήποι που υπάρχουν στα προϊόντα τα οποία αγοράζουν. Και το επόμενο βήμα είναι η απόρριψη των προϊόντων αυτών ώστε να γίνεται η ανακύκλωσή τους και η απόρριψή τους με τον σωστό τρόπο. Η ενημέρωση των καταναλωτών είναι ρόλο και τη Επιτροπή και των κρατών μελών και τώρα έχει τεθεί ε, αυτό το οκταετέ ε, πλαίσιο, το οποίο πιστεύω ότι είναι ακόμη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ. Πάσκα. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στις βιομηχανικές χώρες ο χρόνος ζωής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού συνεχώς περιορίζεται. και βεβαίως ο εξοπλισμός όλο και ταχύτερα ανακυκλώνεται, πράγμα που αποτελεί σοβαρότερο πρόβλημα για το περιβάλλον, συν το χρόνο. Εδώ περιέχονται πολλές επικίνδυνες ουσίες που συχνά δυσκολευόμαστε να απορρίψουμε. Πρέπει καλύτερα να λυθεί το πρόβλημα ήδη από τη φάση του σχεδιασμού των προϊόντων. Καλύτερα να δώσουμε έμφαση την ε, αντικατάσταση των υλικών αυτών από άλλα λιγότερο επικίνδυνα. Το, κυρίως στην περίπτωση του PVC είναι πολύ δύσκολο να τηρηθούν με αυτό το υλικό οι ε, απαιτήσει για περιβαλλοντική προστασία, αλλά δύσκολα ε, αντικαθίσταται αυτό το υλικό. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει εκ νέου η κυρία Δαμανάκη εξ της Επιτροπής, ευχόμενη στον Επίτροπο κύριο Ποτότσνικ ε, ταχύ ανάδοση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε εισηγητά, κυρίε εισηγήτρια, μέλη του Κοινοβουλίου, θέλω να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για τη σκληρή δουλειά της. Χάρη σε αυτή τη σκληρή δουλειά φαίνεται ότι εμφανίζεται συμφωνία διαμορφώνεται συμφωνία στο Κοινοβούλιο. Πράγμα πολύ σημαντικό. Το Κοινοβούλιο δηλαδή, δηλαδή θα διατυπώσει ένα σύνολο κανόνων βάσει των οποίων τα προϊόντα που θα κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά δεν θα περιέχουν κάποιες επικίνδυνες ουσίες. Φυσικά η πρόταση αποτελεί συμβιβασμό. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι συμβιβασμοί οδηγούν σε συμβιβασμούς. Αυτό είναι προφανές. Επίσης είναι προφανές ότι το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και όλοι οι άλλοι έχουν δείξει καλή θέληση και καταλήξαμε σε κάτι που μπορεί η πλειοψηφία μας να το υποστηρίξει. Πολλά έχουμε να πούμε φυσικά εκ μέρους της Κομισιόν. Θέλω να πω ότι θα θέλαμε το, το πεδίο εφαρμογή του συμβιβασμού να είναι περισσότερο σαφές όσον αφορά την εφαρμογή στα κράτη-μέλη και όσον αφορά με τις επιχειρήσεις τη, το, μεταβατική περίοδο των 8 ετών. Έτσι λοιπόν στο κείμενό μας ε, αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο θεωρούμε ότι θα εφαρμοστεί αυτός ο συμβιβασμός και θα θέλαμε τα κείμενα αυτά να μπουν στα πρακτικά κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως ε, το θέμα το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά, τον συμβιβασμό αυτό το παίρνουμε πολύ σοβαρά και θα αρχίσουμε ε, να εργαζόμαστε για την αναθεώρηση της, της ε, οδηγίας καθώς θα τίθεται ενισχύ. Επίσης, οι διατάξεις για την αξιολόγηση συμμόρφωσης και τη σήμανση θα έχουν σοβαρό αποτέλεσμα δεδομένου ότι πρέπει να γνωρίζουμε αν τα προϊόντα συμμορφώνονται και με ποιο τρόπο θα επαληθεύεται αυτή η συμμόρφωση. Κατόπιν όλων αυτών, κυρία Πρόεδρε, δεν φτάσαμε στο τέλος της δουλειάς μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους ε, για την βοήθεια και τις προτάσεις σας. Η Κομισιόν θα τις λάβει υπόψη της. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Η κυρία Εύανς, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, καταρχήν, για τα σχόλιά τους. Από τη συζήτηση αυτή καταλαβαίνει κανείς τις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των πολιτικών ομάδων και τη δύσκολη διαδικασία την οποία αντιμετωπίσαμε. Έχουμε όμως την υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων ε, και ελπίζω ότι την Τετάρτη κατά την ψηφοφορία ε, θα φανεί αυτή η συμφωνία. Χαίρομαι ε, για τη δέσμευση της Επιτροπής για την οδηγία αυτή, διότι το μέλλον της ίδιας αυτής της οδηγίας βρίσκεται σχεδόν αποκλειστικά στα χέρια της Επιτροπής εφόσον ε, υπεψηφιστεί την Τετάρτη. Θα έχουμε τις ε, διαδικασίες ε, στην απόφαση, αλλά η Επιτροπή στο μέλλον θα έχει το ρόλο ε, της επανεξέτασης και γι' αυτό θέλω να ζητήσω από την Επιτροπή να θέσει σε προτεραιότητα της μελλοντική, τη μελλοντική επανεξέταση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα απόβλητα τα οποία δημιουργούν ακόμη κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον. Όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, απόψη, είναι καλύτερη η πρόληψη από τη θεραπεία και υπάρχουν πάρα πολλές ουσίες, πολύ περισσότερες από αυτά τα βαρέα μέταλλα και τους επιβραδ διακινητές φλόγας ε, που ε, περιορίζονται με βάση την τωρινή οδηγία ροζ. και σαφώς υπάρχει ανάγκη για περισσότερους μελλοντικού περιορισμούς. Η συζήτηση αυτή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και την παρακολούθησε ένα ευρύ ακροατήριο και στον κλάδο και στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και πιστεύω ότι στην τελική αυτή συμβαστική λύση καταφέραμε να ανταποκριθούμε στους αρχικούς στόχους της οδηγίας ΡΟΣ και έχουμε τώρα ένα αποτελεσματικό νομοθετικό μέσο εφόσον το ψηφίσει το Κοινοβούλιο την Τετάρτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πέρα ούτε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει Τετάρτη. 12. Προχωράμε με κάποιες ανακοινώσεις.